Ε, η οποία είχε διακοπεί στις 17 Δεκεμβρίου συνεχίζεται. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς το νέο έτος ε, ξεκίνησε παρόμοια με το όπως τελείωσε το προηγούμενο με πολύ βία μετά από τις διαπραγίες στο Παρίσι, στην ε, Τζακάρτα, στη Κωνσταντινούπολη στις 17 Ιανουαρίου στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης έγινε μια βαριά δολοφονική επίθεση και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπεσαν ε, θύματα. Δέκα πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θανατώθηκαν και νέα άλλοι ε, τραυματίστηκαν. Στο Μακατούκο πέθαναν πάνω από δύο ντουζίνες ε, άνθρωποι μετά από μια τρομοκρατική επίθεση την Παρασκευή το βράδυ και υπάρχουν και 15 βαριά τραυματισμένοι. Πραγματικά συμπάσχουμε και πενθούμε με τις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμεθα ε, γρήγορη ανάρρωση. Αλλά δυστυχώ θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι η τρομοκρατία πλέον δεν γνωρίζει σύνορα και θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι στόχο είναι η ελευθερία μα και μα απελεί όλου, είτε στην Τουρκία είτε στο Μπορκίνα Φάσο ή σε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποια άλλη περιοχή του κόσμου. Γι' αυτό κυρίε και κύριοι, ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι μια καθημερινή απειλή η τρομοκρατία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει πραγματικά να κλονιστούμε από αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις, αλλά θα πρέπει να καταβάλουμε την κοινή προσπάθεια να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία στη βάση των δημοκρατικών μας πεπιθήσεων, μέσω της χρήσης της αστυνομίας, ε, της εφαρμογής του κράτους δικαίου, αλλά κυρίως με αύξηση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. νομίζω ότι όλοι πραγματικά σαν βαθιά θλίψη για τα θύματα και τους οικείους τους. Τα πρακτικά και τα αγκριθέντα κείμενα της συνεδρίασης της 17ης Δεκεμβρίου είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν ενστάσεις εδώ. Όχι.